ο ηγέτης του κόμματός μου ε, που τον βάρεναν ε, η ελευθεροτυπία, η ελευθερία του λόγου στην Ολλανδία διαφυλάσσεται πρόεδρος διακόπτη. Τι σχέση έχει αυτό με τις εργασίες μας εδώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Α, έχουμε και γραπτή δήλωση πρώτα απ' όλα. Που συνέλεξε τις απαραίτητες υπογραφές. 14 του 2011 του κυρίου Κωνσταντίνου Πουπάκη Χάουιτ και τα λοιπά και άλλων συναδέλφων για ένα εθελοντικό σύστημα επισήμασης Μπράγε στις συσκευασίε βιομηχανικών προϊόντων έχει συγκεντρώσει πάνω από τα μισά μέλη του Κοινοβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού θα διαβαστεί ε, στους αποδέκτες και θα δημοσιευθεί με τα ονόματα των υπογραφών που θα καταχωρηθούν στα πρακτικά. Ο κύριος Πουπάκης νομίζω ήθελε το λόγο σύντομα σας παρακαλώ.